θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Βάσει του άρθρου 156, οι πρόεδροι των ε, επιτροπών με ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση στη διάσκεψη των ε, πρόεδρων των επιτροπών ως προς τη σύσταση της Επιτροπής Τραν ε, για τη συγκεκριμένη εκτελεστική πράξη. Αν δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση από κάποια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 μέλη εντός 24 εμόρ, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται, αλλιώς θα τεθεί προς ψήφιση.